Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Όπως σας είχα πει και το πρωί, κατά την έναρξη των εργασιών, πρέπει να κάνω κάτι το οποίο δεν έκανα στην περασμένη συνεδρίαση. Να διαβάσω δηλαδή τις αποφάσεις των συντονιστών της προηγούμενης συνεδρίασης, της 16 Σεπτεμβρίου ούτω ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στα πρακτικά και να είναι εκτελεστέ οι αποφάσει. Σε εκείνη λοιπόν τη συνεδρίαση οι συντονιστέ αποφάσισαν για την αποστολή στη Γαλλία. Στο Notre Dame de Lande. Η διάσκεψη των Προέδρων όμως απέρριψε την αποστολή αυτή για διαδικαστικούς λόγους. Και έτσι οι συντονιστές αποφάσισαν να επιμείνουν στο αίτημα. Όταν δηλαδή ξεπεραστούν τα διαδικαστικά να επιμείνουν να γίνει η αποστολή. Για την αποστολή στην Ιρλανδία οι συντονιστές κατέγραψαν την απουσία εκπροσώπων της αντιπροσωπείας που είχαν ζητήσει οι συντονιστές και επομένως υπάρχουν ε, οργανωτικά προβλήματα και γι' αυτό αποφάσισαν να ακυρώσουν την αποστολή στην Ιρλανδία. Προσθέθηκαν επίσης ε, και προβλήματα εκπροσώπησης του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου, ένας λόγος παραπάνω για να ακυρωθεί η αποστολή. Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου, οι συντονιστές αποφάσισαν να εμπιστευτούν τη γραμματεία. Η γραμματεία στις 16 Σεπτεμβρίου είχε κάνει μια πρόταση τροποποίησης με την ενσωμάτωση τεσσάρων σημείων το σημείου για την αξιολόγηση διαχείριση των ε, εργασιών των ε, αναφορών, την οργάνωση δημόσιων ακροάσεων σε συντονισμό με, το, με την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, κοινοβουλευτική επιτροπή, συγγνώμη, και με τη συμμετοχή των συντακτών. Και υπάρχει και ένα τέταρτο σημείο, τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, της ε, οργάνωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το τέταρτο σημείο υπήρξε αρνητική ψήφος από την ε, ομάδα του ΕΛΚΑ. Επομένως αυτό το σημείο δεν ενσωματώθηκε ως πρόταση τροποποίησης του κανονισμού. Και για αυτό το σημείο θα ήθελα να πω στην Κομισιόν ότι η δική μας Επιτροπή θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την παρακολούθηση της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αναπήρων έτσι όπως προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επικυρώθηκε από τον Ιούλιο. Δεν θα τροποποιηθεί λοιπόν ο κανονισμός, αλλά παραμένει ε, ενεργή η συμμετοχή μας ε, ως Κοινοβούλιο, θεσμική συμμετοχή. Οι συντονιστές επίσης το Σεπτέμβριο αποφάσισαν να μην δεχτούν το αίτημα για μία αποστολή μετά από την αναφορά 944 του 2004 για την αδυναμία του, Ευρωπαϊκού, του Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα απόβλητα. Θα γίνουν κάποιες προφορικές ερωτήσεις όμως. Αυτό τον δέχτηκαν για τις απάτες ε, κατά την πώληση εμπορικών προϊόντων και για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην καμπάνια στην Ιταλία. Επίσης, η πρόταση για μια διερευνητική αποστολή στην ε, λεκάνη του ποταμού Εύρου. Ε, απορρίψαμε το αίτημα για ψήφισμα για τη βιώσιμη παραγωγή ε, μελιού. Τελευταίο σημείο των συντονιστών είναι η εφαρμογή, η αποδοχή της γνωμοδότησης νομικής υπηρεσίας για τη διαχείριση των εκθέσεων μετά από τι διερευνητικέ αποστολέ και επισκέψει. Εμεί είχαμε ζητήσει μια γνωμοδότηση νομική υπηρεσία, μετά από την ε, έκθεση που είχαμε συγγράψει για τη Γαλλικία, που δεν βρίσκει σύμφωνο όλου του συμμετέχοντε τη ε, αποστολή. Και η γνωμοδότηση νομική υπηρεσία έπρεπε να καθορίσει μια διαδικασία. Με βάση αυτή τη διαδικασία, το περιγραφικό κομμάτι μια έκθεση, μετά από μια αποστολή, διερευνητική αποστολή, θα πρέπει να είναι καρπός συνεισφορών όλων των μελών της αντιπροσωπείας που αποτελούν την αποστολή. Σε περίπτωση δηλαδή διαφωνίας θα πρέπει να γίνει ένα κείμενο που αντικατοπτρίζει όλες τις απόψεις όλων των συμμετεχόντων στην αποστολή. Στα συμπεράσματα τώρα και στις συστάσεις η νομική υπηρεσία λέει ότι σε περίπτωση που δεν συμφωνούν τα μέλη της αντιπροσωπείας μπορεί να ψηφίσει η Επιτροπή ε, με καθορισμό μιας προθεσμίας για την παρουσίαση τροπολογιών. Σε σχέση λοιπόν με την δική μας περίπτωση, δηλαδή την έκθεση για τη Γαλλικία, ε, αποφασίσαμε να ενσωματώσουμε στην περιγραφή τις απόψεις των τριών μελών της αντιπροσωπείας και να χρησιμοποιήσουμε ως βασικό κείμενο για τα συστάσεις και τις, τα συμπεράσματα, αυτό που θα προτείνει δηλαδή ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας α, και που θα παρουσιαστεί στην συνεδρία του Νοεμβρίου, τις απόψεις αυτές και οι συνάδελφοι θα μπορούν να παρουσιάσουν τροπολογίες που θα ψηφιστούν στην επόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Αυτές είναι οι αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από τους συντονιστές στις 16 Σεπτεμβρίου. Και προφανώς ε, επ' αυτών θα υπάρξει συνένεση από την Επιτροπή, εδώ αναφορών. Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των συντονιστών, σήμερα το πρωί θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Χέφνερ αντικατέστησε τον κύριο Βολεγούκεν, ο αντικαταστάθηκε ο κύριος Σαλαβράκος, ο Μέγερ ε, Κάντι, αντικατέστησε τον κύριο Κάντης και Βαλέζε ο, αντικατέστησε τον Διάρα. Αυτή ήταν οι, αυτές ήταν οι αλλαγές. Πρώτο σημείο, κάποιοι συνάδελφοι ζήτησαν να κλείσει η αναφορά 1298 του 2012, όπως ε, διατυπώθηκε από τον κύριο Πάξας μετά από την προηγούμενη συνεδρία των συντονιστών. Έγινε λοιπόν αυτή η πρόταση και από αυτή της πρότασης οι συνάδελφοι των σοσιαλιστών, των σοσιαλιστών και του Άλντε ζήτησαν να κλείσει ε, σε αντίθεση με το ΕΛΚ ε, και με απουσία της ΓΚΟΕ. Δεν μπορεί να ξανανοίξει όμως η αναφορά λόγω πλειοψηφία. Και μόνο αν υπάρξουν νέα στοιχεία μπορεί να ξανανοίξει αυτή η αναφορά. Έτσι αποφασίστηκε. Σε ό,τι αφορά... Σας παρακαλώ να πάρω το λόγο στο τέλος. Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό, των, την ανάθεση των εκθέσεων των εκθέσεων που θα κάνει η Επιτροπή μας αποφάσισε, μια και οι συντονιστές δεν έχουν άποψη, να χρησιμοποιήσουμε για να αποφασίσουμε τους δύο συγητές τη μέθοδο DONT. Η έκθεση για την Ευρωπαϊκή θα γίνει για το 2013 και η ετήσια έκθεση της Επιτροπής μας για το 2013 πρέπει να καθορίσουμε ποιοι θα είναι οι συντάκτες, οι ε, θα χρησιμοποιήσουμε, όπως σας είπα, τη μέθοδο DON'T. Για τα σημεία C και D. Ετήματα για γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Πρώτον, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το 2014-2020 για την Ιθαγένεια και δεύτερη έκθεση για τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ποια είναι η κατάστασή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ομάδα των συντονιστών αποφάσισε να αντικαταστήσει την γνωμοδότηση και να κάνει ανταυτής γραπτή ανακοίνωση. Για τη συνέχεια που θα δοθεί στην ακρόαση που κάναμε στις 24 Σεπτεμβρίου για την, το αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις της οικονομικής ε, και χρηματοπιστωτικής κρίσης στους Ευρωπαίους πολίτες αποφασίστηκε να ετοιμάσουμε μία ανακοίνωση προς την Επιτροπή ΕΚΟΝ, η οποία έχει ξεκινήσει να συντάσει μία έκθεση με το ίδιο θέμα. Θα είναι μια γνωμοδότηση, όπως σας είπα, θα είναι μια ουσιαστικά υπομορφή ανακοίνωσης που θα περιέχει όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Και όπως ζήτησαν και κάποιοι συνάδελφοι, θα εμπλουτιστεί επίσης και με κάποιες ιδέες για τις επιπτώσεις της κρίσης σε πολίτες που έχουν διάφορες ειδικέ ανάγκες που επηρεάζονται ακόμα πιο σοβαρά από την κρίση από ό,τι οι υπόλοιποι πολίτες. Σε ό,τι αφορά την ατζέντα της Επιτροπής μας για τον Νοέμβριο. Το κείμενο που μοιράστηκε στους συναδέλφους τροποποιήθηκε με την προσθήκη της επίκτρωσης της ε, αναφοράς 847 του 2011 το ζήτησε ο συνάδελφος Βαλέζη και οι συντονιστές ε, δέχτηκαν την ε, συμπερίληψη. Σε ό,τι αφορά το σημείο 4, διαδικασίες και δραστηριότητες της Επιτροπής μας, συζητήσαμε για μια πρόταση κειμένου που παρουσιάστηκε στην Προεδρία από τέσσερις συντονιστές τον κύριο Σαλαβράκο, τον κύριο Βέρτμαν, τον κύριο Μποστινάρου και τον κύριο Γιάρ. Και με τον έγγραφο αυτό οι προαναφερθέντες ε, συντονιστές προβλέπουν ε, διαδικαστικές αλλαγές ούτως ώστε να επιταχύνουμε το, την εξέταση της αναφοράς ούτως ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματική η εργασία μας. Αυτό το έγγραφο εγκρίθηκε από τους συντονιστές με πλειοψηφία. Με την αντίθεση, την κάθετη αντίθεση του κύριου Χέφνερ, ο οποίος αμφισβήτησε και τη μέθοδο και την ουσία και ζήτησε η παρέμβασή του να καταγραφεί στα πρακτικά. Η γραμματεία έδωσε κάποιες, κάποια λεπτομεριακά στοιχεία σημαντικά και θεώρησε ότι αυτό το έγγραφο των συντονιστών είναι θετικό. Και αναγνωρίζεται ομόφωνα η προσπάθεια, η σημαντική προσπάθεια που κάνει η γραμματεία. Κάποια νούμερα που θέλω να σας δώσω. Ε, νούμερα σχετικά με την ε, ανεπάρκεια του προσωπικού στη γραμματεία. Το 2013 η γραμματεία έχασε ένα άτομο. Έχασε μία μονάδα, συγγνώμη, ένα τμήμα. Ε, υπάρχει μια δεύτερη θέση η οποία αντικαταστάθηκε part-time και υπάρχει και μια άλλη θέση η οποία χειρεύει. Ε, Επίση, προέκυψε μια νέα καινή θέση και υπάρχουν και κάποιες θέσεις βοηθητικές που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Δεν είναι επαρκώς επανδρομένη η γραμματεία λοιπόν. Αυτό είναι ανεπαρκές και απαράδεκτο για τους πολίτες και προφανώς είναι και ένας λόγος που καθυστερούμε να απαντούμε στις αναφορές των πολιτών. Επίσης, 500 αιτήσει, λέει η γραμματεία, ε, βρίσκονται σε φάση μετάφρασης. Και μέχρι τον Νοέμβριο, άλλες 275 αναφορές θα υποβληθούν στην Επιτροπή μας προς έγκριση. Αυτό επηρεάζει την ε, αποτελεσματική διεκπαιρέωση των ε, αναφορών. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι από το τέλος του 2012 ε, μέχρι τα μέσα του 2013 είχαμε και πολύ περισσότερες αποστολές και γνωμοδοτήσεις. Επομένως, λογικό είναι να ακολουθηθούν οι κανόνες ε, που προτείνουν οι συντονιστές και να πληρωθούν οι θέσεις που χειρεύουν, τόσο ώστε να απαντάμε πιο γρήγορα στους ε, πολίτες. Επίσης, κάποιες αναφορές είναι επίγουσες. Η 051 του 2013 ε, θεωρήθηκε επίγουσα, τον έκριναν με πλειοψηφία αυτό οι συντονιστές. Δεύτερο αίτημα για χαρακτηρισμό κατεπίγοντος από το Κάρλος Ιτουργκάης ε, αφορά την αναφορά 570 του 2013. Όμως αυτό δεν το δέχτηκαν οι συντονιστές, δεν θεώρησαν ότι πρέπει να χαρακτηριστεί κατεπήγουσα και ζήτησαν να ξεκινήσει ε, μία ε, έρευνα ε, προκειμένου να πληροφορηθούν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τη μοίρα αυτής της αναφοράς. Επίσης, μία άλλη αναφορά, η 1194, η 1713 και άλλη μία του 2013 που ζήτησαν οι συνάδελφοι Παλώνε και Αντζελίλη αυτές θα θεωρηθούν ε, επίγουσες αναφορές. Υπό τα διάφορα, δεχτήκαμε αυτό που μας είπε η κυρία Όκεν, ε, μας το ζήτησε γραπτός. Σας είπα στην αρχή της συνεδρίασης ότι είχε ένα δυστύχημα κυρία Όκεν, γι' αυτό δεν μπορούσε να παραστεί. Ε, καταγράψαμε όμως το αίτημά της να ζητήσει την επικύρωση της σύμβασης του Μαρακές για την ε, χρήση των ε, γραπτών κειμένων από τυφλούς και οι συντονιστές αποφάσισαν να εγκρίνουν ομόφωνα αυτό το αίτημα. Επομένως, θα διατυπώσουμε μια επιστολή προς την Κομισιόν και προς το Συμβούλιο. Υπάρχουν και κάποια ενημερωτικά στοιχεία για τα υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλεί την Επιτροπή ΛΥΠΕ και την Επιτροπή Αναφορών να οργανώσουν ένα εργαστήρι για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Οι συντονιστές επ' αυτού είναι θετικοί. Στο μέλλον λοιπόν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα για την οργάνωση αυτού του workshop. Επίσης ε, ζητήθηκε από την Προεδρία από τους συντονιστές να έρθει σε επαφή με την διάσκεψη των ε, Πρόεδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ούτω ώστε να, να θεωρήσει την απόρριψη του αιτήματό μας για να δοθούν ακόμα δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας. Η Πρόεδρος λοιπόν θα έρθει σε επαφή με τον Πρόεδρο Λένε για να του ζητήσει ακριβώς αυτό το πράγμα. Επίσης σας ενημερώνω όπως αποφάσισαν οι συντονιστές το Σεπτέμβριο η Προεδρία να ετοιμάσει και να υποβάλει κάποια ερωτηματικά, κάποια ερωτήματα, αυτά που ακούστηκαν στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών του Σεπτεμβρίου. Εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα ε, των συνεδριάσεων της Επιτροπής μας για το 2014 και με αυτό τελειώνουμε όλα τα σημεία. Αυτά αποφασίστηκαν. Για το δεύτερο σημείο ο συνάδελφος ζητάει το λόγο, ο συνάδελφος Πάγκου. Köszönöm szépen elnök asszony. Megpróbálok nagyon gyors lenni. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είναι σύντομος. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, σχετικά με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Για παράδειγμα, ε, όσον αφορά την αναφορά 1298 του 2012, η Επιτροπή μας αποφάσισε η αναφορά αυτή να μην κλείσει όσο δεν έχει ε, εκδοθεί απόφαση στην σχετική δικαστική υπόθεση στη Σλοβακία. Πρόκειται λοιπόν για ένα λάθος διαδικαστικό. Οι συντονιστές αποφάσισαν ενάντια στην απόφαση που ήδη έχουν λάβει να κλείσουν την αναφορά αυτή, να ολοκληρώσουν την εξέταση της αναφοράς αυτής. Δυστυχώς, παρότι αρκετοί βουλευτές είπαν ότι δεν θέλουν να κλείσει η υπόθεση. Επιπλέον είναι σημαντικό να δούμε Ε, ε, στον κανονισμό εάν μπορούν οι συντονιστές να κλείσουν ε, αυτή την υπόθεση. Αυτό συνδέεται και με μία αρχή του δικαίου και νομίζω ότι η μειοψηφία έχει λάβει μια απόφαση η οποία δεν αντιστοιχεί στην επιθυμία της πλειοψηφίας. Πιστεύω Μάλλον θα στραφώ προς ε, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου, διότι πιστεύω ότι ε, δεν έχουμε ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία. Ευχαριστώ. Εμπάγκο, καταλαβαίνω την ε, διαφωνία σας, που εν μέρει είναι και δική μου, για να μην πω δική μας. Η πρόθεσή μας είναι πάντα να απαντάμε στους πολίτες που απευθύνονται σε εμάς. Το θέμα είναι αντικείμενο της αναφοράς που συζητήσαμε, που ήταν πάρα πολύ επίμαχη, που συζητήθηκε πολλές φορές. Οι συντονιστές έλαβαν εντολή από την Επιτροπή να αποφασίσουν για αυτό το σημείο, γιατί έγινε αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή και αποφασίσαν να αποφασίσουν τελικά για αυτό το θέμα οι συντονιστές. Να αποφασίσουν οριστικά. Αν τα ερωτήματα δηλαδή που θέτουν οι συντάχτες για να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά είναι βάσιμα. Η πλειοψηφία των συντονιστών, όπως είπα και προηγουμένως, αποφάσισε όμως ότι υπάρχουν επιχειρήματα που επιβάλλουν το κλείσιμο της, της αναφοράς. Κύριε Μπάκο, ξέρετε ότι όταν ένας πολίτης έρχεται για το ίδιο θέμα με νέα στοιχεία, τότε μας ανοίγει τα χέρια. Αν όμως δεν υπάρξουν αυτά τα νέα στοιχεία, ε, δεν μπορούμε να ξανανοίξουμε την ε, αναφορά. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Με βάση τους κανόνες της δημοκρατίας, αποφασίσαμε να διευθυνθούμε με αυτόν τον τρόπο την αναφορά. Οπωσδήποτε εσείς έχετε κάθε δικαίωμα να αναλάβετε να προωθήσετε τις πρωτοβουλίες που αναφέρετε. Κυρία Μπάουερ. Thank you ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που απαντήσατε και στην επιστολή μου παρά τα όσα είπατε, έχω δυσαρεστηθεί που οι, που οι συντονιστές μπόρεσαν ε, ε, να ε, ε, καταργήσουν μια απόφαση της συνεδρίασης της 27ης Μαΐου. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν οι συντονιστές να ακυρώνουν απόφαση της Επιτροπής μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα υποβάλουμε νέα αναφορά στην Επιτροπή μας, εάν αποφασίσετε να κλείσετε την παρούσα, διότι... δεν έχουμε μόνο το θέμα της διπλής υπηκότητας που αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά η διαδικασία αυτή καθ' αυτή δημιουργεί πολύ σημαντική νομική αβεβαιότητα ε, όσον αφορά κάποια βασικά δικαιώματα των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Παρακαλώ. Κύριος Λαζάροφ. Πρόεδρε, θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Με εκπλήσει η απόφαση αυτή στις 27 ε, Μαΐου ήμουν παρόν και το πρώτο λάθος που έγινε είναι ότι οι συντονιστές συζητάνε την υπόθεση αυτή σε κλειστή συνεδρίαση. Μία αναφορά που σχετίζεται με τα δικαιώματα των πολιτών, γιατί είναι κάτι κρυφό. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη λάθος απόφαση και παρακαλώ την Πρόεδρο να σεβαστεί όλους τους κανόνες και τις αρχές μας. Οι προλαλήσαντες αναφέρθηκαν και στο δεύτερο λάθος οι τρεις συντονιστές στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και παρουσία του κ. Κάσκο που δεν είναι καν ε, συντονιστής αυτοί έλαβαν απόφαση στην συνεδρίαση αυτή. Ε, πρόκειται για σημαντικό λάθος. Γιατί δεν ε, αντιμετωπίζουμε σωστά το θέμα αυτό, είναι σοβαρό το θέμα. και ε, είναι ντροπή, όχι απλά λάθο, να εμποδίσουμε έναν υπήκο να ε, λάβει την υπηκότητα άλλη χώρα. Ευχαριστώ όλου όσου πήραν το λόγο. Προσπάθησα να απαντήσω στα email που μου στείλατε. Επαναλαμβάνω ακόμα, μια φορά ότι ο της Επιτροφής μας είχε αποφασίσει να πετάξει το μπαλάκι στους συντονιστές να, για να αποφασίσουν οι συντονιστές. Επομένως έχουν απόλυτη εντολή, έχουν λάβει από την ολομέλεια αυτή την εντολή και άρα δεν υπάρχει καμία παράτυπία. Μπορεί να μην συμφωνείτε. Αλλά εμείς συζητήσαμε επί της ουσίας και τελικά δημιουργήθηκαν δύο στρατόπεδα σε αυτή τη συζήτηση. Αναγκάστηκα να ζητήσουν να ψηφίσουμε σε επίπεδο συντονιστών. Και μετά την ψηφοφορία που έγινε, ελήφθη μια απόφαση. Την απόφαση αυτή σας την κοινοποίησα στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Καταλαβαίνω τη θέση των συναδέλφων που πήραν το λόγο. Αν και νομίζω ότι οι όροι που χρησιμοποίησατε, οι εκφράσει που χρησιμοποίησατε είναι λίγο υπερβολικοί. Δεν υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων κανενό. Δεν υπάρχει καμία, καμία παραβίαση των κοινοβουλευτικών κανόνων, αν μου επιτρέπετε. Αν όμω θεωρείτε ότι κάτι υπάρχει προβληματικό, διορθώσουμε στον τρόπο που εργαζόμαστε, κανένα πρόβλημα να δεχτώ διαταγές και οδηγίες άνωθεν. Κανένα πρόβλημα να διορθώσω τα λάθη που έκανε ενδεχομένω η Προεδρία στη διαδικασία αυτή. Επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά ότι αποφασίζουμε να μην, κρατήσουμε, να μην κρατήσουμε ανοιχτή μια αναφορά περιμένοντας να αποφασίσει μια δικαστική αρχή. Βασικά να μην την κρατήσουμε σε μια εκκρεμή κατάσταση. Έτσι αυτή είναι μια θέση. Επίσημα την κλείσαμε, περιμένοντας νέα στοιχεία. Έτσι, επίσημα την κλείσαμε. Αν υπάρξουν νέα στοιχεία που δικαιολογούν μία συζήτηση ε, ενώπιον ενό οργάνου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα την ανοίξουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η κατάσταση είναι παρκώς ξεκάθαρη και νομίζω ότι και σε άλλες περιπτώσεις αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε πλειοψηφία. Γιατί ακόμα και όταν υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των πολιτών, μερικές φορές ε, δημιουργούνται αντίθετα στρατόπεδα. Τις αντιρρήσεις σας τις εκατέγραψα στα πρακτικά. Τις λαμβάνω υπόψη και μετά τα αυτά κλείνω το σημείο αυτό, κλείνω τις ανακοινώσεις του Προέδρου και εγκρίνουμε τις αποφάσεις, δηλαδή η πλειοψηφία της Επιτροπής κλείνει, ε, εγκρίνει συγγνώμη, αποφάσεις που, πήρε, που πήραν συντονιστές. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το οποίο είναι η αναφορά. Α, εδώ υπάρχει μια αλλαγή. Μια και οι αναφορές οι οποίες υπάρχουν στη ημερησία διάταξη για το απόγευμα, έχουν ένα μόνο υπογράφοντα παρόντα θα δώσουμε με βάση τα ιωθώτα το λόγο σε αυτόν. Θα πάμε λοιπόν στο σημείο 16, ε, αναφορά 660-2011 της Άννα Σπύρα. Η κυρία Σπύρα είναι παρούσα για να μας εξηγήσει αυτή την αναφορά. Πέντε λεφτά έχετε το λόγο. <clears throat> Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί βουλευτές της Επιτροπής Αναφορών, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μου δώσατε σήμερα τη δυνατότητα να σας μιλήσω σε ό,τι αφορά τα πρότυπα ε, γενετικών περιοδικής ε, προστασίας. Ο γιος μου χρειάζεται 24 ώρη φροντίδα, ε, είναι τσαγωνών, ε, χρειάζεται συνεχή φροντίδα και υποφέρει. Πραγματικά πονάω ως μητέρα που βλέπω την κατάστασή του και πραγματικά δεν ξέρω τι θα το συμβεί όταν πεθάνει. Γι' αυτό και αγωνίζομαι για την περιγεννητική περίθραψη στην Πολωνία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα ήθελα να σας πω καταρχάς πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει το άρθρο 35 του χαρτί των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όλοι έχουν ε, το δικαίωμα πρόσβασης ε, στην προληπτική ε, φροντίδα και πρέπει να μπορούν να χαίρουν της προγραμματικής περίθαλψης. Ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης. και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε την παιδική θνησιμότητα. Η UNICEF ε, και τα Ηνωμένα Έθνη το 13 Σεπτεμβρίου παρουσίασαν μια νέα έκθεση βάσει της οποίας το 2012 6,6 εκατομμύρια ε, παιδιά πεθαίνουν καθημερινά ε, κάτω της ηλικίας των 5. Μάλλον πέθαναν το 2012. Όλα αυτά θα μπορούσαμε με πολύ απλά βήματα να τα αποτρέψουμε, ιδίως ό,τι αφορά ε, την ε, τρική φροντίδα για τη μητέρα και για τον νεογνό ιδίως στις πρώτες 24 ώρες της ζωής του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν νέε έρευνες για να, ε, για να δοθεί μεγαλύτερη στην υγεία, την περιγενετική. Αυτά τα λέει η Μάργαρετ Τσάν, η Γενική Διευθύντρια του ε, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Και βέβαια πρέπει ε, να έχουμε υπόψη μας και άλλες δηλώσεις ε, ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις για να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας, όπως λέει ο Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας και συγκεκριμένα στο τμήμα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Εγώ έχω προσπαθήσει από το 2001 έως το 2013 να μου αποδοθεί ε, δικαιοσύνη όταν έγινε γιος μου 14 χρονών ε, μετακόμισα, αναγκάστηκα να φύγω από την Πολωνία ε, το ζήτημά μου συζητήθηκε σε ένα αστικό δικαστήριο και μετά και στον εισαγγελέα υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα, ασφάλματα ένας νευρολόγος που δεν μπόρεσε να πάρει μέρος υπήρξαν καθυστερήσεις τελικά παρήλθε το, παραγράφηκε ε, η όλη ε, ιστορία. Το 2007 δεν μπορούσα να πιθώ σε δικηγόρο, καθυστέρησε υποθεσή μου, υπήρξε κολλησιεργία και συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν όλα και κλεισμένων των θυρών. Η τελική απόφαση δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Κανένα δεν ήθελα να με βοηθήσει δυστυχώ, γι' αυτό και αποφάσισα να αποταθώ εγώ στο δικαστήριο. 27 προσφυγές έκανε, 24 απορρίφθηκαν και εγώ και ο γιος μου χάσαμε, χάσαμε 14 χρόνια ε, μετά από μακρό αγώνα στην Πολωνία για να μας αποδοθεί δικαιοσύνη. Και μάλιστα με όλο το κόστος να το απομιζόμαστε εμείς. Τελευταία 4 χρόνια ζούμε στην Γερμανία. Ακόμα πιο ε, δύσκολο και πολύ ε, πιο δαπανήρες οι όλες οι διαδικασίες. Ούτε καν μπορούσα να πληρώσω το δικηγόρο μου. Και αυτεπαγγέλτος μου ορίστηκε ένας δικηγόρος που όμως δεν παρακολουθούσε την υπόθεση, δεν παρακολουθούσε τη δικογραφία δεν ξέρω αν όλοι λειτουργούν έτσι, αλλά δεν είναι καθόλου σωστό να κλείνουν τα μάτια απέναντι σε πόλη. Γι' αυτό και στρέφομαι σε εσά, στην Επιτροπή Αναφορών, και σα παρακαλώ να προωθήσετε την ασφάλεια, την προστασία των ασθενών με την ε, θέσπιση καλών προτύπων για την περιεντική υγεία, για να μειωθεί η νευνική νησιμότητα και να αποτραπούν ε, πιθανότητες αναπηρίας για τα ε, νεογνά. Η περιεντική φροντίδα, η μείωση της θνησιμότητας είναι στοιχειώδη το να μπορεί να γεννά μια γυναίκα με ασφάλεια να φέρει σε πέρα στην εγκυμοσύνη της η η περιγεννητική φροντίδα και η φροντίδα είναι στοιχειώδη πράγματα. Κάθε γυναίκα επίσης πρέπει να ενημερώνεται, να γνωρίζει τα δικαιώματά της ε, και τις υποχρεώσει όσων πρέπει να τη φροντίζουν. Πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό εγχειρίδιο που να τα αναφέρει αυτά. Επίσης όλες οι υποθέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και θα πρέπει να έχουμε πανευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλεια ό,τι αφορά την τροφαρμακευτική περίθαλψη στι σχέσει μεταξύ των ασθενών, των παρόχων ε, ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών. Και να εκπαιδεύονται, να καταρτίζονται οι επαγγελματίε του κλάδου. Θα ήταν καλό να υπάρχει μια νέα νομοθεσία που θα προστατεύει όλε τι εγγύου, γυναίκε και τα νεογνά, ώστε να έχουμε πανευρωπαϊκά πρότυπα, ιατρικά πρότυπα και διαδικασίε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχει μια κατάσταση όπου ο καθένας κάνει ό,τι του κατεβαίνει. Υπάρχουν ε, ε, κάποιες απαρχαιωμένες πρακτικές, ε, κάποιες ρουτίνες που πρέπει να τις... Ε, ε να, πάψουν πλέον να ισχύουν. Οι γιατροί έχουν ευθύνες, έχουν ε, Επομένως ε, θα πρέπει να μπορούν και να ε, αναλαμβάνουν τις ευθύνες των πραξιών τους ή των σφαλμάτων τους. Και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια σφάλματα στην Πενιντική Φροντίδα γιατί υπάρχουν αδυναμίες. Μόνο ε, στις σκανδιναβικές ε, χώρες, δεν ξέρω έχουμε κάποια στοιχεία εκεί, δεν ξέρω πόσα παιδιά όμως πεθαίνουν ή πόσα νεογνά πεθαίνουν λόγω ακριβώς αυτών των αδυναμιών και κενών. Επίσης, για ένα πρόωρο ε, βρέφος χρειάζονται 10 ε, φορές παραπάνω πόροι για να φροντίσει κανείς ένα τέτοιο πρόωρο ε, παιδί σε σχέση με ένα παιδί που γεννήθηκε στην ώρα του. και βοήθεια πρέπει να βελτιωθεί στην Ευρώπη. Τα χρήματα πρέπει να φροντίσουμε να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν να καταλάβουν την κατάσταση. Οι γονείς μπορούν να καταλάβουν που παλεύουν μόνοι τους και κάποιες φορές δεν γνωρίζουν καν ποια είναι τα πρότυπα στην περιοχική βοήθεια, ε, φροντίδα. Και κάποιοι ε, επαγγελματίε δεν βοηθούν, ε, δεν δείχνουν προθυμία, πεθαίνουν νεογνά. αυτό δεν πρέπει να το δεχθούμε. Όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν το δικαίωμα να ε, γεννήσουν υγιή παιδιά, να ξεκινήσουν τα παιδιά τους στη ζωή όλα από ε, το ίδιο επίπεδο. Εκπαίδευση των γιατρών επίσης. Καλύτερα πρότυπα ε, γενετικής φροντίδας. Αυτά είναι τα βασικά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από πλευράς ε, Επιτροπής μας, η Ζαμπέλ Τελαμάτα. Επιτροπής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνουμε την ε, κατάσταση που παρουσίασε η ομιλήτρια η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με το θέμα της ε, περιγεννητικής υγείας Γνωρίζετε ότι οι νομικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι περιορισμένες στον τομέα της υγείας. Όσον αφορά λοιπόν την περιγεννητική υγεία, μόνο συστάσεις και υποστηρικτικές δράσεις ε, είναι δυνατόν να γίνουν. Στον τομέα της πληροφόρησης για την υγεία δραστηριοποιούμαστε. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε είναι έκθεση περιγεντικής υγείας στην Ευρώπη. Ε, ασχολούμαστε λοιπόν με το θέμα της εγκεφαλικής ε, παραλυσίας και να συλλέξουμε σχετικά στοιχεία. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ομάδες επιρρογνωμόνων ε, στον τομέα της περιγενετικής υγείας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να, να βελτιώσουν την κατάσταση στις χώρες τους. Είναι όμως εθνική αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να οργανώσουν το, σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας τους. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει η Επιτροπή είναι να στηρίξει τα κράτη-μέλη, να στηρίξει τους εμπειρογνώμονες, να στηρίξουμε με προγράμματα και με ερευνητικά προγράμματα. Για παράδειγμα, μόλις έχουμε ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα για μια ευρωπαϊκή στρατηγική και επίσης έχουμε δημιουργήσει ε, ε, ε, μια βάση δεδομένων για, την, για τις έρευνες για την υγεία των παιδιών στην Ευρώπη. Επίσης, η κυρία Σπύρα ανέφερε την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στην υγεία. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να στηρίξει με τα διαρθρωτικά ταμεία την ανάπτυξη καλών στρατηγικών καλών πρακτικών ε, στην υγεία. Όσον αφορά την ε, προώθηση της υγείας και της ασφάλειας, έχουμε μια πρωτοβουλία για την ασφάλεια των ασθενών ε, που τρέχει εδώ και κάποια χρόνια και τώρα με την νέα διασυνοριακή οδηγία που θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε επιπλέον ένα μέσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλουν δείκτες. Είπατε ότι μόνο κάποια κράτη-μέλη υποβάλλουν αναφορά σχετικά με γιατρικά λάθη. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ε, υπολογίζουμε όλα τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Έτσι μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη μας και να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των παιδιών. Όσον αφορά την ε, κατάρτιση των ε, επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, είναι πάλι εθνική αρμοδιότητα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει μέσω διαφόρων προγραμμάτων ε, και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για παράδειγμα. Συνοψίζοντας, προσπαθούμε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη Προσπαθούμε να στηρίξουμε ανάλογα με τις δυνατότητές μας, ε, αλλά δεν είναι δυνατόν να έχουμε ε, απολύτως ενία προσέγγιση, δεν αποτελεί αρμοδιότητα των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαι καν βέβαιη αν είναι αρμοδιότητα των κρατικών αρχών, διότι σε κάποια κράτη-μέλη είναι περιφερειακή αρμοδιότητα η υγεία. Προσπαθούμε πάντως να παρέχουμε όσο γίνεται καλύτερη, καλύτερες υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω λόγο στον κύριο Βαλές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία της, ε, την αναφέρουσα. Από ό,τι άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αυτό λέει η Επιτροπή ουσιαστικά. Έχω μια ερώτηση τι δικαιώματα, τι υποχρεώσεις θα πρέπει να έχουν οι γυναίκες όταν ε, γεννιέται το παιδί τους. Δεν θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι έχουν όλες οι γυναίκες τα ίδια δικαιώματα τις ίδιες υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως ε, του που λαμβάνει χώρα ο τοκετός και ανεξαρτήτως του που μένει η γυναίκα. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό φυλάδιο, ενημερωτικό φυλάδι, μια μελέτη για, την, ε, για τον ασφαλή τοκετό. Ένα τέτοιο εγχείριο θα μπορούσε να υπάρχει. Και γιατί πιστεύετε ότι τελικά τα λάθη ε, συγκαλύπτονται ή τέλος πάντων κανείς δεν αντλεί ε, διδάγματα από αυτή την ε, κατάσταση. όχι δεν μπορείτε να έχετε αναφέρει στο το λόγο, θα δώσω τώρα στον κύριο Μποστινάρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω. Τη μία βέβαια την, προλα... την ανέφερε ο συνάδελφος Προβαλέσα που μίλησε πριν. Πρώτο ερώτημα, πώς ορίζεται αυτό που λέμε ε, το κετό υγιή γένα και πρότυπα. Ε. Όλα αυτά πρέπει να είναι ενιαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια στο εσωτερικό των χωρών. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με τι πρακτικέ σε κάθε χρόνο, γιατί μιλάμε και για τι ιατρικέ πρακτικέ που ισχύουν σε κάθε χώρα και για την εκπαίδευση. Πώ θα δημιουργήσουμε μια ομοιομορφία και ποια νομικά πρότυπα, ποιου νομικού κανόνε θα δημιουργήσουμε. Εγώ έρχομαι από μια ορθόδοξη, κατάγομαι από μια ορθόδοξη χώρα, ξέρω ότι όλοι έχουμε υποχρεώσει και όλοι έχουμε δικαιώματα. Πώς ορίζουμε το μεν, πώς ορίζουμε το δε και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τις εφαρμόζει τις υποχρεώσεις αυτές, αν υπάρξει κάποιο σφάλμα. Δεύτερο ερώτημα. Εκφράστε την άποψη ότι κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν καμιά ανάλυση, καμιά αξιολόγηση της υγιούς του υγιούς πακέτου, όπως το είπατε εσείς. Και όταν γνωρίζουμε ότι το σύστημα υγείας είναι επικουρικότητα εν γέννη. Πώ θα δεχθείτε ή θα θέλετε να επιβληθούν ευρωπαϊκά πρότυπα, γιατί είναι αυτό σε αντίθεση με τι συνθήκε τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Και αν μετά να πω και κάτι άλλο. το να φέρει μια γυναίκα στον κόσμο ένα παιδί είναι και μια προσωπική ευθύνη, προσωπική τεράστια προσωπική ευθύνη για τους ώμους μιας γυναίκας, μιας οικογένειας. Και κάποιες φορές δεν είναι και οι δύο γονείς, ε, αλλά και ο πατέρας έχει ευθύνε και η μητέρα. Πολλές οικογένειε ε, είναι μονογονεϊκές. Πώς αυτή την ευθύνη τεράστια μπορεί κανεί να την μεταφέρει σε ένα θεσμό που είναι μακριά και απομονωμένος. Είναι δυνατόν να δουλέψει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Θα μπορούσε κάποιο στις Βρυξέλλε να αποφασίζει τι συνιστά έναν ε, υγιή τοκετό και ότι εφαρμόστηκαν σωστά τα πρότυπα και να αποφασίζει δυνητικά ότι πρέπει να κινηθεί δικασία παραβάση για παραλήψεις ή για σφάλματα σε κάποια χώρα. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ρωτήθηκαν αρκετά από τους προαλήσαντες συνάδελφους. Δεν θέλω να κάνω ρωτήσεις γιατί εσείς οι έρθατε εδώ γιατί νιώθετε βοήθητοι. Και έτσι συνήθω νιώθουν οι αναφέροντες όταν έρχονται σε εμά, γιατί έχουν εξαντλήσει κάθε οποιοδήποτε άλλο ε, οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο ή άλλο τρόπο είχαν στη χώρα τους και γι' αυτό έρχονται εδώ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μόνο που θέλω να ξέρω είναι το εξής. Έχετε πραγματικά εξαντλήσει όλα τα εθνικά ένδικα μέσα που ήταν στη διάθεσή σας. Γιατί είστε εδώ σήμερα, γιατί είστε εδώ τώρα. Είστε εδώ γιατί έληξαν πλέον, τερματίστηκαν όλες οι... όλα τα διαβήματα που κάνουν σε εθνικό επίπεδο και δεν μπορεί να γίνει τίποτα πια εκεί. Δεν είναι θέμα εθνικής ε, οργάνωσης υγείας, εθνικού συστήματος υγείας. Από την άλλη πλευρά, κοινωνικές πρωτοβουλίες στη βάση δεν βοηθάνε αυτά. Δεν βοηθάνε τις γυναίκες. Γιατί υπάρχουν. Η εντύπωση που αποκόμισα εγώ προσωπικά από τη δική σας αναφορά είναι ότι θέλετε να απευθύνετε ε, μια έκκληση να ε, αντιμετωπίζονται, να, να ε, υπάρχει καλύτερη μεταχείριση για αντιμετώπιση των γυναικών ιδιών αυτών που κυοφορούν. Ακούστηκαν πολλές ερωτήσεις που απευθύνονται προς την ε, συντάκτρια της ε, αναφοράς. Θα ήθελα να απαντήσει αν το επιθυμεί. Με το μικρόφωνο παρακαλώ. Φυσικά θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ευτήρων, όπου συμμετέχουν 36 χώρες, έχει καθορίσει κάποια πρότυπα τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται και στις 36 αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να λειτουργούμε. Υπάρχει αυτό το πλαίσιο, αλλά κάθε ατομικό κράτος μέλος θα αποφασίσει τι πρότυπα θα, θα εφαρμόσει. Έχουμε πιο φτωχές χώρες, πιο πλούσιες χώρες, ε, εγώ τα τελευταία χρόνια ζω στη Γερμανία και προφανώς τα πράγματα ως προς την ιατροφαρμακευτική υπερήθαλψη είναι τελείως διαφορετικά από την Πολωνία. Υπάρχουν κάποια συστημικά λάθη που παρατήρησα στην Πολωνία και τα οποία δεν υπάρχουν στη Γερμανία και χρειάζεται χρόνος για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι θύμα του συστήματος και δεν θα ήθελα κάποιο άλλο να περάσει την τραυματική αυτή εμπειρία που πέρασα εγώ τα τελευταία χρόνια τα τελευταία 14 χρόνια. Ε, λόγω του ότι είναι τμήμα ενός ε, λανθασμένου συστήματος. Όταν μιλάω, μιλάω ως μητέρα. Κοιτάω γύρω μου και βλέπω ότι... και έχω την αίσθηση ότι μόνο οι γονείς ε, αντιδρούν με τέτοιον τρόπο. Φυσικά υπάρχουν μητέρες οι οποίες είναι θύματα, υπάρχουν παιδιά τα οποία πέθαναν, ε, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες... Ε, πρέπει να φροντίσουν 24 ώρες το 24 το παιδί τους και δεν θα μπορέσουν να έρθουν εδώ να σας μιλήσουν. Εγώ αυτό που θέλω είναι να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει αυτό το πλαίσιο το οποίο το πλαίσιο προτύπων που σας εφάρμοσα, που σας συγγνώμη, ανέφερα. Ε, μιλάμε για ποιοτικά πρότυπα, για μια δέσμη καλών νέων προτύπων που πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν πρέπει να σκορπίζουμε τα χρήματα των φορολογουμένων μας, ούτως ώστε να πεθαίνουν τα παιδιά μας. Πρέπει να επενδυθούν χρήματα τους ώστε να καταπολεμήσουμε την ε, παιδική θνησιμότητα και τα, την αναπηρία. Είπα και το ξαναλέω ότι οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να γνωρίζουν τις ευθύνες και τα δικαιώματά τους. Σας μίλησα για αυτόν τον οδηγό για τις εγκύους γυναίκες. Το 50% ε, των εγκυμοσύνων στην Ευρώπη δεν είναι προσχεδιασμένες συχνά η έγκυος γυναίκα δεν ξέρει τι πρότυπα ισχύουν. Φερρυπίν, τι είδου ε, τεστ πρέπει να κάνει, τι είδου εξετάσει πρέπει να κάνουν, ειδικά σε πιο φτωχέ χώρε. Προσπαθούν να κάνουν εξοικονόμηση χρημάτων. Στην Πολωνία, Φερρυπίν, βρισκόμαστε πολύ, ε, πολύ από το σωστό μοντέλο που θα έπρεπε να εφαρμόζεται. Ε, μία γυναίκα, ας πούμε, ε, συνήθως δεν μπορεί να πάει σε δημόσια νοσοκομεία, αλλά πρέπει να πάει σε ιδιώτη γιατρό. Και δεν μπορεί κάθε φορά να πληρώνει αυτά τα λεφτά και όλε οι γυναίκε κατά ανάγκη. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα οδηγό που να λέει τι εξετάσει πρέπει να κάνει, ποιε εξετάσει είναι υποχρεωτικέ, τι δικαιώματα έχει, τι υποχρεώσει έχει, όταν πάει στο νοσοκομείο για να γεννήσει, α πούμε, τι δικαιώματα έχει. Όλα αυτά σα τα λέω από πρώτο χέρι, από εμπειρία. Υπάρχουν πολύ καλοί γιατροί, όντω, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι γιατροί όσο σκληρά και να δουλεύουν, είναι άνθρωποι και μπορεί να κουραστούν και αυτοί κάποια στιγμή. Μερικέ φορέ δουλεύουν ατελείωτε ώρε. Αν πίν. Πάρουμε το παράδειγμα μιας, ενός χειρουργείου, ε, όπου γεννάει μια γυναίκα. Τι εξοπλισμό πρέπει να έχει αυτό το χειρουργείο για τον τοκετό. Πόσες ώρες ε, μπορούμε να αφήσουμε μια έγκυο γυναίκα έτοιμο να γεννήσει χωρίς γιατρό. Την αφήνουμε εκεί στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου χωρίς γιατρό. Εγώ πέρασα μια ολόκληρη μέρα χωρίς να με δει κανένα. Εγώ έκανα ό,τι έπρεπε να κάνει. Εγώ πήγαινα στο γυναικολόγο μου. Έκανα όλες τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνω. Άρα και αυτές οι υποχρεώσεις πρέπει να αναφέρονται στον οδηγό. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ελέγχει, να ξαναελέγχει πού πηγαίνουν τα λεφτά. Ξοδεύονται σωστά τα λεφτά. Γιατί το Ευρωπαϊκό αυτό Συμβούλιο ε, με ευτήρων και γυναικολόγων ε, εξόδευσε τόσο πολύ χρόνο για να δημιουργήσει αυτά τα πρότυπα, τα οποία εμείς τα αγνοούμε και δεν τα εφαρμόζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι πραγματικά εφαρμόζονται. Φυσικά, σαν μητέρα σας μιλάω, αλλά την απόφαση εσείς θα την πάρετε. Η περιγεννητική περίθαλψη είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί 500.000 ε, παιδιά γεννιούνται πρόωρα είναι ένα τεράστιο κίνδυνο για την Ευρώπη. Αν αυτά τα παιδιά ε, έχουν ε, κάποιο πρόβλημα, κάποια αναπηρία, ποιο θα τα φροντίσει. Κανένα άλλο δεν θέλει να πάρει τον λόγο. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πρόταση. Θέλετε να κρατήσουμε από ό,τι καταλαβαίνω ότι αναφορά ανοιχτή και να περιμένουμε μια διαφορετική απάντηση. Ο κ. Μποστινάρου. Πρόεδρε, ίσως θα ήταν σοφό να διαβιβάσουμε την αναφορά αυτή στην Επιτροπή Υγείας ε, για να έχουμε και τη δική τους αξιολόγηση και να δούμε με δικά τους μάτια, με τις δικές τους ε, ε, αρμοδιότητες σε την κατάσταση, διότι η τραγωδία αυτή είναι πραγματική. Πρόκειται για μια τελείως οριακή κατάσταση. Είναι πολύ σοβαρή. Για να οριστούν λοιπόν ε, σωστά τα λάθη με κοινού Ευρωπαϊκού όρους, αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε στο μέλλον κάποιες από τις ε, τραγικές αυτές περιπτώσεις, τις οποίες αναφέρθηκε η αναφέρουσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Να παραπέμψουμε την αναφορά στην Επιτροπή Δημόσιας Υγείας. Μ' αρέσει εμένα η πρόταση του κυρίου Αποστινάρο και αναρωτιέμαι αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Μπορούμε να διαβάσουμε την αναφορά σε άλλη επιτροπή και να στήσουμε γνωμοδότηση. Αν μπορούμε, τότε θα συμφωνήσω απολύτως με τον κύριο Ποστινάρο. Συμφωνώ κι εγώ. Χρήσιμο θα ήταν να απευθύνουμε ένα τέτοιο αίτημα προς την ε, καθήλυνα αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Όμως η συνθήκη, την οποία επικαλέστηκε και ο κ. Μποστινάρου, μας δίνει ακόμη μια άλλη δυνατότητα. Γιατί στο άρθρο 178, στην παράγραφο 5, η συνθήκη μιλάει για το δρόμο που μπορεί να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να κάνει μια παρέμβαση, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε το θέμα στο Συμβούλιο, να ακούσουμε την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή των Περιφερειών, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο στόχο τη συνθήκη, δηλαδή το υψηλό επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ειδικέ ειδικά περιπτώσει, εξασφαλίζεται. Μπορώ αυτή την περίπτωση να την θεωρήσω ειδική περίπτωση, γιατί τα νούμερα που μας έδωσε η συντάκτρια είναι πραγματικά ανησυχητικά. Και νομίζω ότι θα τιμήσουμε και στη, τη συνθήκη, αν εμείς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή και επομένως ως Κοινοβούλιο, μια και εκπροσωπούμε το Κοινοβούλιο, ζητήσουμε την εφαρμογή μιας διάταξης ε, της συνθήκης που μιλάει για το δικαίωμα στη ζωή και την προστασία της ζωής. Ούτως ώστε μετά από μία συζήτηση να ψηφίσουμε για να ζητήσουμε περισσότερα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ούτως ώστε να προωθήσουμε τη διακοπή της εγκυμοσύνης. Το θέμα της ζωής, το θέμα της γέννησης, το θέμα της προστασίας της υγείας, αυτών των θεμελιωδών αξιών είναι πιο σημαντικά από αυτά που προσπαθεί τώρα να, προωθήσει, να προωθήσουν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και από τις αρμόδιες εθνικές αρχές να πάρουν θέση. Θα μπορούσαμε να, ζητήσουμε, να στείλουμε μία επιστολή, ούτως ώστε να ζητήσουμε επιβεβαίωση των αριθμητικών στοιχείων που λάβαμε ή άρνηση ότι ισχύουν. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, και άλλα στοιχεία και άλλες απόψεις. Να μην ακούσουμε μόνο μία άποψη, αλλά να ακούσουμε και τη γνώμη της, ε, του επίσημου πολωνικού κράτους. Σίγουρα θα στείλω το θέμα αυτό στην ε, Επιτροπή Δημόσιας Υγείας. Θα ζητήσω επίσης να γίνει μια μελέτη, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 178 της Συνθήκης και θα στείλω, όπως σας είπα, και μια επιστολή στην πολωνική κυβέρνηση για να πει τη θέση της για τα όσα ακούσαμε σήμερα. Αν συμφωνείτε επίσης, παραμένει ανοιχτή η αναφορά αυτή. Ευχαριστώ τη συντάκτρια, την κυρία Σπύρα. Και πάμε στην επόμενη αναφορά. Βασικά είχαμε αλλάξει τα σημεία της ημερήσιας διάταξης και πάμε πίσω. Θα πάμε στην αναφορά 1454 του 2012 του Γίλιαμ Σάντερς, Βρετανικής Ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις εις βάρος Άγγλων φοιτητών στη Σκοτία, όσον αφορά την καταβολή των διδάκτρων. Ο συντάκτης δεν είναι δεν είναι παρόν, θα δώσω το λόγο στον Αντώνιο Μάρκο. Ευχαριστώ πολύ. Το πρόβλημα με αυτή την αναφορά είναι ότι σύμφωνα με τον Ετούντα ε, γίνονται διακρίσεις εις βάρος ε, Άγγλων ε, σπουδαστών στα σκοτσέζικα πανεπιστήμια, διότι τα σκοτσέζικα πανεπιστήμια τους χρεώνουν υψηλότερα δίδακτρα από ό,τι από άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να αναφέρει κυρίως ότι είναι εσωτερικό θέμα από νομικής πλευράς, δεδομένου ότι ε, οι διακρίσεις αφορούν μόνο εγχώριους φοιτητές, Ουαλούς, Σκοτσέζους, Άγγλους ε, και Βόρειους Ιρλανδούς. Πρόκειται λοιπόν κυρίως για διάκριση μεταξύ αυτών των φοιτητών ε, κάτι που δεν συνδέεται καθόλου με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τέτοιες υποθέσεις πρέπει να ε, αντιμετωπίζονται σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θεωρεί ότι ε, οι αρχές και τα δικαστήρια της Μεγάλης Βρετανίας είναι αποκλειστικά αρμόδια για την περίπτωση αυτή. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Μία σύντομη ερώτηση. Υποθέτω ότι είναι σωστή η απάντηση της ε, Κομισιόν, αλλά ε, αντίκειται στο αίσθημα δικαίου των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε οι πολίτες να αναπτύξουν ευρωπαϊκό αίσθημα ταυτότητας ε, ε, δεν πρόκειται... Ε, πρόκειται σαφώς για υπόθεση διακρίσεων, διότι γίνεται διάκριση ανάμεσα στους εγχώριους και τους αλλοταπούς. Δεν θα πρέπει λοιπόν τουλάχιστον το κράτος μέλος να αιτιολογήσει τέτοιες διακρίσεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Πράγματι δεν μας αφορά εμένα. Ε, το αίσθημά μου είναι όπως για παράδειγμα στη Γερμανία που μιλάμε για τα διόδια, εάν πρέπει να πληρωθούν διόδια θα πρέπει να τα πληρώνουν όλοι. Ε, δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι μόνο οι αλλοδαποί πληρώνουν διόδια. Μήπως είναι πράγματι περίπτωση ε, διακρίσεων, διότι γίνεται διάκριση με βάση την καταγωγή. Ή έχω καταλάβει κάτι λάθος, γιατί δηλαδή απορρίπτεται την ε, αναφορά αυτή. Thank um, Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει στην απάντησή της ότι πράγματι πρόκειται περί διάκρισης. Αλλά είναι διάκριση μεταξύ ε, εγχωρίων φοιτητών, ε, δεν γίνεται η διάκριση λόγω υπηκότητας, διότι όλοι αυτοί οι φοιτητές, ε, Άγγλοι, Σκοτσέζοι, Ουαλοί και Ιρλανδοί, είναι Βρετανοί. Και σε αυτή τη φάση το δικαστήριο δεν έχει θεωρήσει ότι αυτό είναι κάτι που εμπίπτει στο ευρωπαϊκό δίκαιο και θεωρεί ότι είναι εσωτερικό θέμα. Δεν εφαρμόζεται δηλαδή εδώ ευρωπαϊκός νόμος. Αλλά οι πολίτες αυτοί μπορούν να προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια και να παρουσιάσουν την κατάσταση αυτή. Δεν είναι αβοήθητη δηλαδή. Ευχαριστώ. Ο Φερνάντο. λαμπίτια. Κάπως έτσι. Αυτό να προσπαθήσετε, Πρόεδρε, να προφέρετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι περίπλοκο το θέμα. Είχα και εγώ ένα γιο που σπούδαζε στο Μπάρτ στην Αγγλία. υπάρχει ένα σύστημα ανεξαρτήτως του που σπουδάζει κανείς, ε, το ίντερ και τα λοιπά, αλλά έχουμε ε, με τη Σκοτία και τη Βρετανία δύο διαφορετικές ε, κυβερνήσεις με τις ποσοστώσεις έχουν, αποφασίζουν Λονδία, στην Βρετανία να τριπλασιάσουν τα διδακτρά αλλά διατηρούν τα σκοτσέζικα πανεπιστήμια τα δίδακτρά του σε επίπεδο που τα έχουν. Και γι' αυτό υπάρχει εισβολή κατά κάποιο τρόπο ε, Βρετανών φοιτητών προ τα ε, ε, σκοτσέζικα πανεπιστήμια γιατί πληρώνουν τρεις φορές λιγότερα δίδακτρα. Τι αμυντικού μηχανισμού μπορεί να ε, θεσπίσει η κυβέρνηση τη σκοτία. Όταν ανεβαίνουν τρεις φορές τα διδακτρά στην, τι να κάνει στην Βρετανία, να κάνει το ίδιο. Δεν θα ήταν αυτό καλή ε, πολιτική. Διότι με αυτό που έκανε η Βρετανική κυβέρνηση οδήγησε σε κύμα φυγής φοιτητών προς τα σκοτσέσικα πανεπιστήμια. Τι μπορεί να κάνει το σκοτσέσικη κυβέρνηση. Αν ήταν ανεξάρτητο έθνος και κράτος η Σκωτία δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχουν οι Σκοτσέζοι είναι ότι δεν είναι ούτε Γερμανοί, ούτε Μαλτέζοι, αλλά Σκοτσέζοι που είναι υπήκοοι του Βασιλείου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά έχουν δικαίωμα να προασπίσουν ε, τις πολιτικές ό,τι αφορά τι ποσοστώσει, ε, τα δίδακτρα και αυτό που καλό είναι, ε, καλό είναι να κάνουμε είναι να πληρώνουν οι φοιτητέ από την Αγγλία, ε, την Ουαλία και τη Βόρεια Ολλανδία αυτά που πληρώνουν στην πατρίδα του όταν έρχονται στη Σκοτία. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να κάνει. Καταλαβαίνω σε τι θέση βρισκόμαστε. Είναι δύσκολη η θέση μα. Δεν μπορούμε να πιέσουμε ούτε καν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αντικειμενικά. Είναι καταφανής διάκριση αυτή για λόγους που δεν θέλω να σχολιάσω τώρα, αλλά συμβαίνει στο εσωτερικό μιας χώρας. Άρα εδώ σταματάει η πρωτοβουλία που μπορεί να πάρει ή οι πρωτοβουλίε που μπορεί να πάρει η οι Επιτροπή. Παραμένει πάντως μία περίπτωση καταφανούς διάκρισης εις βάρος κάποιων Ευρωπαίων πολιτών δεν τους εξασφαλίζει το δικαίωμά τους στην κινητικότητα, που είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δίδακτρα που πληρώνουν κάποιοι ε, είναι πολύ ψηλότερα από τα δίδακτρα που πληρώνουν στο ίδιο πανεπιστήμιο κάποιοι άλλοι. Επειδή εδώ μεταξύ στη χώρα τους αυτοί οι άνθρωποι ε, είναι, έχουν πολύ ψηλά δίδακτρα, ε, έχουν πρόβλημα να, να μείνουν εκεί. Από την άλλη υπάρχει πρόβλημα κινητικότητας. Μπορεί να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσε όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει σε επαφή με τις εθνικές αρχές, να έρθει σε επαφή, ας πούμε, ε, με τον αρμόδιο Υπουργό Παιδεία, για να μάθει για ποιου λόγους υπάρχει αυτή η στάση στη χώρα αυτή. Μόνο και μόνο για να υπάρξει μια κάποια θεσμική συνεργασία. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να παρεύουμε στα εσωτερικά μια χώρα, γιατί όπω υπόθηκε δεν έχουμε ειδική αρμοδιότητα να μπούμε στην ουσία ενό τέτοιου θέματο εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνάδελφο Φερνάντο θέλει ξανά το λόγο, παρακαλώ. Δεν είναι ότι διαφωνώ μαζί σα, κυρία Πρόεδρε. Αλλά με την κολοκυθιά εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να να μείνουμε στι ποσοστώσει. Έχουμε, ε, παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση του γιού μου που σπουδάζει στο Μπαθ, στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία και πληρώνει τριπλάσια δέκτρα από ό,τι θα πλήρωνε στη χώρα των Βάσκων ή μπορεί να πληρώσει δέκα φορέ παραπάνω άμα ε, αυξηθούν τα δέκτρα. Δεν είναι το πρόβλημα Σκοτίας, Βρετανίας. Ή θα βάλουμε ε, παντού τις ίδιες ε, ε ποσοστώσεις. 9.000 πληρώνει κάποιος αγγλικές λίρες ε, και 100 ευρώ στη, χώρα των Βάσκων φοιτητής. Και στην Ισπανία τα διαφορετικά πανεπιστήμια έχουν διαφορετικά δίδακτρα ανάλογα με την ε, αυτόνομη περιφέρεια. Θέλουμε να υπάρχει κινητικότητα φοιτητών και σπουδαστών. Εάν θέλουμε τότε θα πρέπει ε, να είναι οι τιμές, ε, όπως και για τη βενζίνη θα μπορούσαμε να πούμε, ότι OK, για να υπάρχει κινητικότητα θα βάλουμε την ίδια τιμή της βενζίνης παντού. Μα δεν είναι αυτό όμως η λύση. Yeah. Also ich habe das schon äh, Νομίζω ότι δεν ε, θα πρέπει να μπλεχτούμε στο ύψος των ε, διδάκτρων των πανεπιστημίων. Τα πράγματα έχουν ως έχουν. Ε, μπορεί κάποιος να διαφημίζει ότι έχει χαμηλά διδακτρά, άλλοι διαφημίζουν ότι έχουν πολύ ψηλά. Έπασε τόση. Αυτό, σε αυτό δεν μπλεκόμαστε. Αλλά ε, λέμε ότι ένας Σκοτσέζος πληρώνει χ ε, δίδακτρα, ένας Γερμανός πληρώνει τα ίδια, ενώ ένας Άγγλος πληρώνει υψηλότερα. Εγώ απλά ήθελα να προσθέσω ότι Πολύ σωστό θα είναι η Κομισιόν να ε, χρησιμοποιήσει τα κανάλια επικοινωνίας ε, που έχει. Υπάρχει λοιπόν η Επιτροπή Αναφορών, υπάρχει και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Ε, θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι αγαπητό Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα. Ε, εγώ ε, θα το παρέπεμπα αυτό στους αρμόδιους, διότι είναι εσωτερική υπόθεση κράτους μέλους. Ε, προφανώς δεν μπορούμε να πλεχτούμε σε αυτό. Από την άλλη παραμένει μια περίπτωση διακρίσεων. Ευχαριστώ. Η πρότασή μου είναι μειονοτική, όπως βλέπω. Δεν υποστηρίζεται. Θα πρέπει να κλείσει λοιπόν αυτή η αναφορά και να διαβιβαστεί στην αρμόδια ε, Εθνική Επιτροπή, μας τον αρμόδιο φορέα, που είναι η Επιτροπή Αναφορών του Ηνωμένου Βασιλείου. Κλείνουμε λοιπόν την αναφορά του σημείου 14. Πάμε στο σημείο 15 του Μάικλ Κέιν, Βρετανός πολίτης, Αναφορά 1186 του Μάικλ Κέιν, Βρετανική Ιθαγένεια, σχετικά με την ε, ιατροφαρμακευτική κάλυψη Βρετανών πολιτών που διαμένουν στη Γαλλία και την αναφορά 1218 του 2007 του Πίτερ Τζοβτζεύσκη, ε, η Βρετανική Ιθαγένεια, σχετικά με την ε, ιατροφαρμακευτική κάλυψη Βρετανών πολιτών που διαμένουν στη Γαλλία. Ε, δίνω το λόγο κατευθείαν στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν είναι παρόντε οι συντάκτε αναφορά. Thank you very uh, much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ παλιά αναφορά. Ξεκίνησε το 2007. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε ε, μια σειρά από καταγγελίες από οικονομικά ανενεργά άτομα που ζούσαν στη Γαλλία και είχαν δυσκολία στο να αποκτήσουν πρόσβαση στην καθολική ιατρική περίθαλψη. Κινήθηκε τη δικασία επιβολής κυρώσεων κατά της Γαλλίας, γιατί θεώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αντιβαίνει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο η Γαλλική νομοθεσία. Συναντηθήκαμε πολλές φορές με τις γαλλικές αρχές και το 2011 έκαναν μια, ένα νέο νομοσχέδιο, κυκλοφόρησε μια νέα εγκύκλιο. Δεν συμφώνησε η Κομισιόν με κάποια σημεία αυτή, τη μελετήσαμε πάντως. Και γι' αυτό και δεν σταματήσαμε τη διαδικασία αυτή επιβολή κυρώσεων. Επίση, στο μεταξύ λάβαμε και άλλε καταγγελίε. Μετά από συναντήσεις με τους Γάλλους αποφασίστηκε η δημιουργία ενός ε, σημείου πρόσβασης όπου ξένοι αλλοδαποί πολίτες που κατοικούν στη Γαλλία και που δεν έχουν ε, πρόσβαση στο ΣΕΜΗ μπορούν να πάνε σε αυτό το σημείο πρόσβασης που κατά περίπτωση εξετάζει τα αιτήματά τους. Τον Ιούνιο του 2013, φέτος συστάθηκε αυτό το κέντρο, κάποιες υποθέσεις ε, μάθαμε ότι επιλήθηκαν, κάποιες άλλες όχι. Η θέση της Κομισιόν λοιπόν είναι ότι η διαδικασία αυτή πολύ κυρώσεων παραμένει ε, σε εκκρεμότητα, την κρατάμε μέχρι να έχουν επιληθεί όλες οι υποθέσεις και μέχρι ό,τι λάβουμε επιβεβαίωση από τις γαλλικές αρχές. Γκάιθ. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κάποιος το λόγο. Είπατε ότι ζητήθηκα περισσότερες πληροφορίες. Μας τα είχατε πει ε, και τα είπατε και στη γαλλική κυβέρνηση, άρα παραμένει ανοιχτό ο διάλογος. Επομένως, θα περιμένουμε την ανακοίνωση να δούμε τι θα λέει και μετά θα τοποθετηθούμε για το κατά πόσο θα αφήσουμε ανοιχτή και θα κλείσουμε την αναφορά αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, στο περθόν 16 μέρες μη δυνατότητα διαβίβαση στην Πολωνία δικαστικών και εξωδίκων εγγράφων προ επίδοση και κοινοποίηση μέσω συμβατικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρόμη. Η αναφορά 277 και υπάρχει και δεύτερη αναφορά ε, η 1399 και οι δύο από πολλούς υπηκόους. Η δεύτερη αναφορά είναι σχετικά με την ελληπή δυνατότητα στην Πολωνία για επίδοση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων. Πρόσφυγες Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, και οι δύο αναφορέ που έλεξαν την προσοχή τη Κομισιόν στην ε, ελληνική εφαρμογή τη ε, νομοθεσία του 2007 σε ό,τι αφορά την ε, επίδοση δοκιμάτων, ε, εγγράφων δικαστικών και εξοδίκων και για την ερχόμενη παραβία στο άρθρο 18 συγγνώμη, της συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολωνίας. Δύο, με δύο άρθρα του πολωνικού κώδικα αστικής δικονομίας αναλύσαμε. Το πρώτο επιβάλλει υποχρέωση στις πλευρές ε, μιας εμπορικής ε, ε, υπόθεσης όταν κατοικούν στην Αλοδαπή να ορίσουν έναν πληρεξούσιο νομικό εκπρόσωπο για την επίδοση αυτών των εγγράφων στην Πολωνία. Αν δεν οριστεί όμως ένα τέτοιο πρόσωπο, τα έγγραφα τα οποία απευθύνονται ε, στον διάδικο αυτών κατατίθεται στο δικαστήριο και εκεί μετά επιδίδονται στο διάδικο. Το άλλο θέμα αφορά ένα άρθρο του κώδικα της ε, αστικής δικονομίας ε, της Πολωνίας που λέει ότι η ημερομηνία επίδοση ενός εγγράφου είναι η ημερομηνία της ε, αποστολής της ε, στο δικαστήριο ή η σφραγιδα του ταχυδρομείου. Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση ορισμού ενός ε, πληρεξουσίου νομικού προσώπου, αντικλήτου στην Πολωνία, αυτό το εξέτασε στο δικαστήριο πρόσφατα κιόλας σε υπόθεση Άλντερ 325 11 η ετοιμιγωρία έγινε γνωστά Δεκέμβριο του 2012. Και ποια είναι η ετοιμιγωρία του δικαστηρίου. Το δικαστήριο καταλήγει ότι όταν παραλήψει του εγγράφου κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, η επίδοση ενός δικαστικού εγγράφου πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού για την επίδοση εγγράφου. Επομένως, Ένα σύστημα το οποίο απαιτεί ορισμό αντικλήτου με την επίδοση ενός εγγράφου σε έναν άνθρωπο που διαμένει σε άλλο κράτος δεν συνάδει με τον κανονισμό αυτό. Σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα, κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υποχρέωση να δοθούν τα έγγραφα μόνο σε ένα πολωνικό ταχυδρομικό φορέα σε αντίθεση με το άρθρο 18, διότι συνιστά διακριτική μεταχείριση υπέρ του πολωνικού ταχυδρομικού φορέα. Άρα συνιστά έμεση διαχείριση, ε, διακριτική μεταχείριση για λόγους εθνικότητας, λόγω εθνικότητας. Σε συνέχεια όλων αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τι πολωνικές αρχές για το θέμα αυτό ήδη από το 2011 και τέλος το 2013 οι πολωνικές αρχές μας κοινοποίησαν ότι τα δύο άρθρα άλλαξαν τα εν λόγω του κώδικα πολιτικής οικονομίας, πολιτικής οικονομίας και ήδη έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Πολωνίας 2 Αυγούστου του 2013 ημερομηνία δημοσίευσής τους. Επομένως, για τις αστικές υποθέσεις στην Πολωνία πλέον δεν είναι υποχρεωτικό ένας διάδικος που διαμένει σε άλλο κράτος μέλος να ορίσει πρόσωπο για την επίδοση των εγγράφων. σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα, οποιαδήποτε άλλη ε, πάροχη, οποιαδήποτε πάροχη ταχυδρομικών υπηρεσιών και όχι μόνο οι πολωνικοί μπορούν να αναλάβουν να εκτελέσουν αυτή την επίδοση. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πια συνάδουν ε, οι διατάξεις του πολωνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έκλεισε η Κομισιόν το φάκελο, για μας δηλαδή πλέον είναι λήξαν το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο θέλει το λόγο, κύριε Γιάρ, παρακαλώ. <clears throat> Σύντομη διευκρινιστική ερώτηση. Η Κομισιόν όταν λέει ότι έχει λυθεί το θέμα, τότε η ερώτησή μου είναι αυτό βοηθάει του αναφέροντες ή υπάρχουν προβλήματα μεταφορά στο δίκαιο, προβλήματα εφαρμογής. Καταλάβατε την ερώτηση. Να την ε, διατυπώσει πάλι ο κύριος Γιάννη. Ξαναρωτώ. Η Κομισιόν είπε ότι γενικά αναγνωρίζεται το πρόβλημα και λέει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί επίσης. Θεωρητικά. Αλλά έχει λυθεί έτσι το πρόβλημα και για τον αναφέροντα. Λαμβάνει ηλεκτρονικά τώρα ε, τα έγγραφα. Εάν έχει λυθεί το πρόβλημα και για τον αναφέροντα, τότε μπορούμε να κλείσουμε την ε, αναφορά. Εάν όμως πούμε ότι ωραία εντάξει ε, ενημερωθήκαμε αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα, αυτή είναι η ερώτησή μου. Μισό λεπτό. Θα δώσω τον λόγο στην εκπρόσωπο της Κομισιόν αλλά και εγώ κύριε Γιάρ κατάλαβα, έτσι νομίζω τουλάχιστον, με ναι, βάλει και τα κουστά να με καταλαβαίνετε, ότι με, την, ε, ε, με τις επαφές που είχε η Κομισιόν με την πολωνική πλευρά ε, διευθετήθηκε το θέμα, έγινε κατανοητό το πρόβλημα. Δεν ξέρω, μπορεί να μας απαντήσει την ερώτηση για η Επιτροπή για να αποφασίσουμε και εμείς τα κάνουμε την αναφορά. Ε, well, in the opinion of the Commission... κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να κλείσει η αναφορά γιατί δεν υπάρχουν άλλα εφαρμοστικά μέτρα. Οι δύο διατάξεις του αστυνομικού κώδικα που ήταν κατά του, μάλλον έχοντας αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν υφίστανται πλέον γιατί με τη νέα εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημεία της ε, πολιτικής κυβέρνηση τον Αύγουστο αντικαταστάθηκαν, άρα λύθηκε το πρόβλημα. Πρόεδρο, πολύ ωραία. Αν είναι έτσι τα πράγματα και έτσι τα ερμηνεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Τελευταίο υπό τι είναι η αναφορά 18 δηλαδή μάλλον το σημείο 18 αναφορά 1691 από τον Έρβιν Μικαέλε, Γερμανική ηθαγένεια, σχετικά με τη σύνταξή του από την Ιταλία και τον Ιταλικό Συνταξιοδοτικό Φορέα η NPS. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην περίπτωση αυτή θα έλεγα ότι η αναστολή ε, μιας σύνταξης από την ε, εταιρεία INPS ε, δεν βασίζεται σε ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ουσιαστικά ε, προβλέπει την συνέχιση των πληρωμών ε, σύνταξης αναπηρίας από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο, ακόμα και σε περίπτωση που έχει γίνει μετατροπή μιας σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γύρατος. οι πληροφορίες που έχουμε δεν αρκούν για να μπορούμε να καθορίσουμε εάν έχει παραβιαστεί το, εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο από ε, τον φορέα INPS. Γι' αυτό καλούμε τον ε, αναφέροντα ε, είτε να εξετάσει το θέμα σε εθνικό επίπεδο ή να έρθει σε επικοινωνία με το Solvit και θα πρέπει να δώσει και τον προσωπικό αριθμό ασφάλισής του για να μπορέσει να γίνει εντοπισμός του φακέλου του. Κοιτάξτε, αν όμω αυτό έρχεται, μα τα βοήθεια και τον γυρίζουμε πίσω στη χώρα του, του λέμε λάθο κάνατε από την Ιταλία να αναζητήσετε, τι προφορές δεν ξέρω, μήπως υπάρχει κάποια άλλα φόρμουλα. Να οδηγήσουμε αυτόν τον πολίτη κάπου διαφορετικά. Στο Σόλβιτ θα του λέγαμε εμείς από όλες κομισιόν να απευθυνθεί με βάση πληροφορίε τις οποίες έδωσε στην Επιτροπή Αναφορών. Δεν μπορούμε να πούμε αν παραγνωρίστηκε και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θέλαμε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες. Τον συμβουλεύουμε να απευθυνθεί στο Solvit για να ρυθμιστεί υπόθεσή του με βάση την εθνική νομοθεσία. Παρακαλώ, μπείτε. Ναι, θα πρότεινα, θα πρότεινα να το ανακοινώσουμε αυτό στον ε, αναφέροντα. Βλέπω ότι υπάρχουν δύο προβλήματα. Δηλαδή, πρώτον, θα πρέπει να του πούμε να απευθυνθεί στο Solvit και δεύτερον, μπορούμε επίσης να του πούμε ότι λόγω έλλειψης πληροφοριών ε, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ε, αν έχει γίνει παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Ζητάμε δηλαδή περισσότερες πληροφορίες αν έχει. Προτείνουμε λοιπόν να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Το βασικό πρόβλημα φαίνεται να είναι ότι ο, φορέας, ε, ο στασιωτικός φορέας INPS δεν επικοινωνεί καθόλου ε, με τον αναφέροντα, το οποίο είναι <laughs> απίστευτη αγένεια. Θα πρέπει τουλάχιστον να συνομιλούν μαζί του. Δεν έχει ενημερωθεί γιατί, σταμάτησαν, ε, σταμάτησε η καταβολή της συνταξής του. Να τον καλέσουμε δηλαδή να ε, στραφεί στο INPS ε, και αν έχει περισσότερες πληροφορίες και θεωρεί ότι έχει ε, γίνει παραβίαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου να μας ενημερώσει. Νομίζω ότι συμφωνεί και η Κομισιόν με αυτό. Εγώ θα έκανα άλλη πρόταση, Πέτερ, σε σχέση με αυτό που λες, για να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Θα μπορούσαμε εμείς να γράψουμε στον οργανισμό ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα, και να μην πούμε αυτό στον αναφέροντα, γιατί θα μείνει στη λιάλη τους κακομίδης, κατάλαβες. Λοιπόν, να γράψουμε στον οργανισμό εμείς ως επιτροπή αναφορών για αυτό το θέμα και να μας δώσει ο οργανισμός μια απάντηση για αυτό το θέμα. Και εμείς θα ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λάβουμε την απόφασή μας. Συμφωνείτε, ωραία. Δεν υπάρχουν άλλα σημεία στη μεσιά διάταξη σε ό,τι αφορά το σκέλος Α και σε ό,τι αφορά το σκέλος Β, όπως πάντα. Βάσει τι απαντήσει που δόθηκαν ε, στην Επιτροπή με βάση άλλα έγγραφα μπορούμε να τι θεωρήσουμε ότι έχουν κλείσει. Αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα ή καταγγελία θα διαβιβαστούν τα σχετικά στη γραμματεία, η οποία θα ε, λάβει την Και Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Κλείνω τη συνεδρίαση τη Επιτροπή Αναφορών. Α, όχι. Όχι. Βιάστηκα. Υπάρχουν τέσσερα σημεία. Τέσσερις αναφορές από το σκέλος Β για να μείνουν ανοιχτές έχουμε αιτήματα. Το 36 είναι το πρώτο. το guide. 390, και 390. Sobre el grupo de peticiones και σε ό,τι αφορά ε, τις ε, αναφορές για τον Ευρωπαϊκή Θαγένεια. Κύριε Σντανόκα, που δεν έβλεπα καλά τέλος πάντων, ναι, κύριε Στανόκα μας ζητάει να αφήσουμε τέσσερα σημεία, 66, 65, 67, να τα αφήσουμε. Δεν διαβάζω και καλά τα νούμερα. Δεν μπορείτε να μας τα πείτε τα νούμερα, καλύτερα εσείς, γιατί δεν... Ποιο είναι το... 42. 42 είναι το τελευταίο. Όχι, όχι. Για την Ιθαγένεια 63. Τι είναι το αριθμό, θέλετε. 1444, 1445, 1461, 1542. Όλα από το 2012. Και η 1298. Πάλι για τη διπλή ποιότητα. και το Jugendamt. ...979. Πρόεδρος, ναι, το βλέπω, το βλέπω τώρα. Ναι, μας είχατε στείλει και κάποια άλλα σημεία. Άρχισα εγώ από το τρίτο, αλλά είχατε και άλλα δύο πιο πριν. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Ωραία προσθέτω και αυτό το σημείο και τα δίνω όλα στη γραμματεία. Οπότε τώρα πλέον μπορώ να κλείσω την συνεδρία. Σε ευχαριστώ. Συγγνώμη, δεν την ε, περαίωσα ακόμα τη συνεδρία. Θέλει να πει κάτι ο κύριο Γιάρ. Ναι. Για τα πρακτικά θέλω να φέρω. Νομίζω ότι με αρκετά χαλαρό τρόπο ξανανοίγουμε αυτές τις αναφορές. Μήπως θα το συζητήσουμε. Αν κάποιο θέλει να ξανανοίξει μία αναφορά, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Πρέπει να ακουστούν νέα επιχειρήματα μέσα σε δύο μήνε για το κατά πόσο θα πρέπει να ανοίξει αυτή η αναφορά και να γίνει μια συζήτηση. Να καταγραφεί λοιπόν στα πρακτικά η γνώμη μου είναι ότι ανοίγουμε με πολύ μεγάλη χαλαρότητα και άνεση αυτές τις αναφορές ξανά. Δεν θέλω συνέχεια να ανοίγουν και να κλείνουν αναφορέ έτσι. Πρόεδρε, καλό είναι να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα με μια κάποια διαδικασία. Γιατί αν κάποιο όντω ε, έχει ένα πρόβλημα, να ξανανοίξει αναφορά. Εντάξει, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, συμφωνούμε απόλυτα. Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα άλλο, κυρία μου. Ελπίζω τώρα πια να μην υπάρχουν άλλε ερωτήσει και όντω να κλείσαμε. Θεωρώ λοιπόν ότι κλείνει η σημερινή συνεδρίαση. So Mark, what about this?